και από τις 9 ως τις 12 το βράδυ. Η εμερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας και σας εύχομαι καλή νύχτα.